ακυρώνεται. Η ακόλουθη γραπτή δήλωση έχει υπογραφεί από Ευρωβουλευτές η παριθμόν 32 του 2012 για το Ευρωπαϊκό Έτος για την συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της επαγγελματικής ζωής. Χάρκιν, Μόρε Σαρτιέ, Αντζελίλη, Γιούτα Στάινμπρουκ. Με τα ονόματα των προσυπογραφώντων θα ενταχθεί στα πρακτικά τη συνεδρίαση και έτσι θα δημοσιευθεί. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει ένα, μια διόρθωση όσον αφορά την 6η ε, Φεβρουαρίου 2013 στο κείμενο που εγκρίθηκε.